Dear colleagues, please attention, we will start with... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε με την ε, κοινή μας συνεδρίαση. Παόλο, θα μιλήσω ισπανικά. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργίας σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Μια κοινή συνεδρίαση λοιπόν της Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Γυναικών η οποία λαμβάνει χώρο για να ανταλλάξουμε απόψεις για την έκθεση σχετικά με τις γυναίκες και τον ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές. Είναι ένα σημαντικό θέμα και οι δύο επιτροπές επιθυμούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ζωής των γυναικών των αγροτικών περιοχών. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η κοινή συνεδρίαση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πολλές αγροτικές περιοχές έχουν προβλήματα δημογραφικού χαρακτήρα, προβλήματα εγκατάλειψης των περιοχών αυτών Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πόσο σημαντικό είναι να το συζητήσουμε τώρα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη των δύο επιτροπών και πιστεύω πως πρέπει να αρχίσουμε χωρίς καθυστέρηση και να δώσουμε το λόγο στις δύο συνεισηγήτριες. Στην κυρία Πετήρ, καταρχάς, η συγγήτρια της Επιτροπής Γυναικών. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάσω σήμερα την έκθεση για τις γυναίκες και το ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές. Θα χαρώ λοιπόν πολύ να ακούσω τις απόψεις σας και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όσους συνεργάστηκαν, τις και οδείς και οι τα μέλη της Επιτροπής και τη Γραμματεία η ζωή των γυναικών στις αγροτικές περιοχές διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ωστόσο, πολλές φορές οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές δεν έχουν επαρκή κοινωνικό ε, ιστό, επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες έτσι ώστε να ζουν καλά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε παρατηρήσει πολλούς νέους, πολλές νέες γυναίκες να εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμογή τη αγροτικής μας πολιτικής και αυξάνει τους κινδύνους οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο και από αυτές μόνο το 30% διοικείται από γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε μέσα από το Ταμείο ε, Γεωργικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Πέθρου και να τα ε, διοχετεύσουμε στην ε, βελτίωση της ζωής γυναικών. Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα, ακολουθούν διάφορες ε, και διαφορετικές μάλλον ζωές, πολλές φορές ο ρόλος τους είναι αόρατος και αυτό φαίνεται και στην κοινωνική τους θέση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε πως τα κράτη-μέλη πρέπει να υλοποιήσουν στο έπακρο την υφιστάμενη νομοθεσία έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις και η άνηση μεταχείριση σε βάρος των γυναικών. Οι γυναίκες στην Ήπεθρο έχουν ένα πολυδιάστατο ρόλο ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων, με την προστασία του περιβάλλοντος, με την οικογένεια και η συνεισφορά των γυναικών πρέπει να αναγνωριστεί. Πρέπει να αναγνωριστεί διότι οι γυναίκες συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Και είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να παρέχουν όλα τα ε, δυνατά μέσα στις γυναίκες της υπαίθρου, να, να αντλήσουν κονδύλια από όλα τα ε, διαθέσιμα ταμεία έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και εργασίας των γυναικών, να βελτιωθεί πρόσβαση στην εκπαίδευση, η χορήγηση ε, δανείων στις γυναίκες επιχειρηματίες και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες ε, να παραμείνουν στην Ήπεθρο, να βοηθήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη έτσι ώστε να συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα υψής της ποιότητας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν και για πολλούς άλλους λόγους είναι πολύ σημαντικό να ε, βελτιώσουμε την θέση των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πετήρ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία κυρία στη συζητήτρια της Επιτροπής Γεωργίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω Όσου συνεργάστηκαν μαζί μου στη σύνταξη αυτή τη έκθεση. Και θα ήθελα να εστιάσω στα δικαιώματα των γυναικών και στις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών στην Ήπεθρο. Τώρα, όταν λέμε Ήπεθρο, αγροτικές περιοχές, τι εννοούμε. Ε, πολλά και διάφορα. Υπάρχουν γυναίκες που ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα, ανάλογα το που βρίσκονται, ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα με διαφορετικές οικονομίες. Οικονομίες όμως που χαρακτηρίζονται κυρίως από τη γεωργική δραστηριότητα. Τα δικαιώματα λοιπόν των γυναικών αγροτών δεν ε, είναι πλήρως αναγνωρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν και πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ε, το εξής πρόβλημα. Μία γυναίκα αγρότης που ε, ασχολείται με την, την οικογενειακή επιχείρηση δεν, γίνεται, ε, δεν αναγνωρίζεται ως ε, επαγγελματίας. Υπάρχουν μάλιστα πολλές περιπτώσεις όπου οι γυναίκες δεν έχουν καμία απολύτως προστασία. Για παράδειγμα, σε μια οικογενειακή γεωγική εκμετάλλευση, μια γυναίκα που δεν έχει στην νόμιμη κατοχή της ε, την γη δεν έχει και κανένα δικαίωμα στην ε, επιχείρηση. Πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ούτε στην παραγωγή ούτε και στι ε, πληρωμές, Ακριβώ γιατί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στη γη. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οικογενειακές, δύσκολες διαζύγια, ε, στα κληρονομικά θέματα πολλές φορές ε, ε, μένει κανείς μετά από μια ολόκληρη ζωή στη δουλειά χωρίς τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα στην έκθεση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την ανάγκη να προχωρήσουμε στα πλαίσια των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων την προώθηση της γυναίκας των δικαιωμάτων ανδρών γυναικών που έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες φυσικά υποχρεώσεις. Να σχολιάσω επίσης το τι σημαίνει να καλύπτεται κανείς από τα θέματα της κοινωνικής ασφάλειας στον γεωργικό τομέα. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες η συμπερίληψη στην κοινωνική πρόνοια διαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν ενταχθεί αλλά με πάρα πολύ μεγάλη κατηστέρηση διότι δεν θεωρούνται ιδιοκτήτριες ή εργαζόμενες και έχουμε επίσης και πάρα πολύ ε, σημαντικές διαφορές εξ αυτού και στο ύψος των συντάξεων για τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα. Αυτό που μας απασχολεί επίσης είναι ότι σχετικά και με την κρίση συναντάμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στην κοινωνική ασφάλιση. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να συμπεριλάβουμε εδώ κάποιες προτάσεις έτσι ώστε να μπορεί κανείς ανάλογα με τη συμμετοχή και τα έσοδα της επιχείρησης να συμπεριλαμβάνεται στην κοινωνική ασφάλιση. Ένα άλλο θέμα που αφορά τις γυναίκες στην Ήπεθρο είναι οι δημόσιες υπηρεσίες. Ε, η κάλυψη των αναγκών σαν παράδειγμα των ηλικιωμένων. Στην ουσία είναι κάτι το οποίο θεωρείται ε, η φροντίδα των παιδιών, η φροντίδα των ηλικιωμένων, υποχρέωση των γυναικών. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν ε, οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες που θα μπορούσαν να στηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν οι υπηρεσίες αυτές να αντιμετωπίζουν και την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για στήριξη των γυναικών που υφίστανται την ανδρική βία και επίσης ε, ε, να υπάρξουν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα εργαστούν στον τομέα της πρόληψης ε, της άσκησης βίας εις βάρος των γυναικών από πλευράς των ανδρών. Νομίζω λοιπόν ότι ο χώρος που έχουμε μπροστά μας θα πρέπει να εμπλουτιστεί έτσι ώστε να έχουμε μία πρόταση η οποία να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη για την κατάσταση των γυναικών που ασχολούνται με τη γεωργία ή που κατοικούν σε γεωργικές περιοχές. Ευχαριστώ κυρία Σέρνα. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τους σκιώδεις εισηγητές και των δύο επιτροπών. Έραντς Γκαρθία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τις δύο εισηγήτρες για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχουν κάνει. Μιλάμε για δύο διαφορετικές ε, επιτροπές, ε, την Επιτροπή Γεωργίας και την Επιτροπή ε, Γυναικών από την άλλη. Παρ' όλα αυτά υπήρξε πολύ καλή συνεργασία σε ορισμένους τομείς σαν παράδειγμα η βελτίωση των δυνατοτήτων και των μέσων αναγνώρισης της εργασίας που παρέχουν οι γυναίκες. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε επίσης τις υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν την εργασιακή ζωή και την οικογενειακή ζωή της γυναίκας, ιδιαίτερα σε, σε, περιοχές της υπαίθρου, που είναι η κατάσταση πολύ πιο περίπλοκη από τις αστικές περιοχές και γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερη έξοδος των γυναικών από τις γεωργικές περιοχές και λιγότερο των ανδρών. Ακριβώς αυτό δείχνει τις δυσκολίες της επιπλέον που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον γεωργικό κόσμο. Θα πρέπει να υπάρξει επίσης μια αναφορά στις ενώσεις των γυναικών όχι μόνο ε, για να δούμε με τι ασχολούνται οι γυναίκες αλλά για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να καταλάβει ότι ε, αν δεν εργάζονταν οι γυναίκες με τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν η κατάσταση στον γεωργικό κόσμο θα ήταν πολύ χειρότερη. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν κοινωνική αναγνώριση της υπηρεσίας των γυναικών. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να στηρίζουν την εργασία των γυναικών. Ε, θα πρέπει να ανοίξουν οι αγορές. Μια γυναίκα ας πούμε η οποία έχει ένα κατάστημα, ένα εμπορικό κατάστημα θα πρέπει να θεωρείται εφόσον είναι ιδιοκτήτρια της συγκεκριμένη επιχείρησης ότι θα πρέπει να έχει πλήρη δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών. Και επίσης θα πρέπει ε, να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες και στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου και ιδιαίτερα και της ε, χωροτακτικής ανάπτυξης. Creo que eh, la titularidad compartida de las explotaciones, como ha eh, ε, Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει ε, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εφόσον σε ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες δεν έχουν από κοινού ιδιοκτησία και δικαιώματα, αδικούνται ουσιαστικά θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε σε όλα τα κράτη-μέλη να προσφερθούν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις προς τις γυναίκες. Θα πρέπει επίσης να ευνοηθεί η κατάρτιση των νέων και κυρίως των γυναικών, γιατί οι σωστά εκπαιδευμένες γυναίκες σε έναν τομέα όπως ο γεωργικός κόσμος θα είναι σε θέση να μην λειτουργούν παρά, αλλά και να μην λειτουργούν απλά για τον εαυτό τους, αλλά να στηρίζουν επίσης και τη γεωργία και την κτηνοτροφία στην οποία ενεργοποιούνται και άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν οι οποίες ε, συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης του γεωργικού τουρισμού ε, θα πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι οι άνδρες. Και θα πρέπει επίσης να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην πίστοση και στην μικροπίστοση στις γυναίκες οι οποίες αναλαμβάνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο γεωργικό κόσμο. Έτσι θα δραστηριοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις γυναίκες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να συγχαρώ ακόμα μία φορά τις δύο εισηγήτριες. Ευχαριστώ κυρία Ράντς. Η κυρία Βίφριντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τις δύο εισηγήτριες για την δουλειά την οποία έκαναν, σημαντική σε δύο ε, τομείς, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Η μία πλευρά είναι αυτή η οποία συνδέεται με τις ε, επιχειρηματίες γυναίκες στον τομέα της γεωργίας, γυναίκες που αποκτούν, αγοράζουν, κληρονομούν μια γεωργική δραστηριότητα και την διαχειρίζονται λόγω οικογενειακών λόγων, γυναίκες ε, γεωργών, κόρες ε, γυναικών, αγεωργών, συγγνώμη, ή και κάποιες άλλες γυναίκες οι οποίες για λόγους επιχειρηματικότητας και αν, ακόμα και αν δεν έχουν γεωργικές καταγωγές ασχολούνται με θέματα της γεωργίας σε περιοχές της υπαίθρου. Υπάρχουν επίση και γυναίκες που ασχολούνται με τη γεωργία ε, στα πλαίσια μιας γεωργικής οικογένειας, οι οποίες δεν έχουν καθορισμένο ρόλο, τον οποίο όμως η προσφορά είναι καθοριστική για την επιβίωση της επιχείρησης. Αναφέρθηκαν σε αυτά με διάφορους τρόπους οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν. Ιδιαίτερα για αυτή τη δεύτερη κατηγορία η πρόταση είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Θα ήθελα να επιμείνω ακόμα περισσότερο και για το πρώτο κομμάτι. Φυσικά και συμφωνώ με το κείμενο, αλλά εγώ θα ήθελα να βοηθήσω ακριβώς την ολοκλήρωση της συμμετοχής των γυναικών και της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ήπεθρο και όχι μόνο το προστασίας των γυναικών που εργάζονται στη Γεωργία. Το να δούμε τις γυναίκες μόνο μέσω της προσφοράς τους σε σχέση με την συμμετοχή τους σε οικογενειακές δραστηριότητες είναι περιοριστικό. Ε, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευράς ε, των κρατών μελών. Μία θα έλεγα καταγραφή των γυναικών που ασχολούνται με τη γεωργία και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και σε επίπεδο εργασίας είναι προϋπόθεση. Θα πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα προς τα πίσω, διότι αν στόχος είναι πραγματικά η, η, η η ανάδειξη των αοράτων γυναικών της γεωργίας έτσι ώστε να αποκτήσουν συγκεκριμένα πλέον δικαιώματα, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η κατάρτιση. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών σε μαθήματα για τη γεωργία και σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει σημασία λοιπόν τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την συμμετοχή αυτή, να προωθήσουν ακριβώς την επαγγελματικοποίηση σε εισαγωγικά της θέσης των γυναικών στην γεωργία, έτσι ώστε να είναι μια συνειδητή επιλογή και όχι ένας τομέας ο οποίος επιβάλλεται ή αυτοεπιβάλλεται λόγω της οικογενειακής καταβολής. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αποκτήσουν την αξιοπρέπειά τους, να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να παίξουν σημαντικό ρόλο. Η λεγόμενη ροζ γεωργία είναι πιο αηφόρα και πιο φιλοπεριβαλλοντική. Γι' αυτό ακριβώς η γενική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να της δοθούν κίνητρα και να υπάρξουν γυναίκες σε θέσεις διαχειριστικές. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης και ό,τι έχει σχέση με την ιδιοκτησία της επιχείρησης, την πρόσβαση στην πίστοση, την διαλειτουργικότητα και άλλους τομείς του οποίους οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διευκολυνθούν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρυνθούν έτσι ώστε να πάρουν μέτρα που να ανταποκρίνονται στο πλαίσιο το οποίο έχουν ανάγκη. Και όπως υπογράμμισαν οι συγχύτριες θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και τα δικαιώματα τα κοινωνικά των γεωργών, των γυναικών γεωργών που δραστηριοποιούνται χωρίς να αναγνωρίζονται από πουθενά πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος τους και να υπάρξει πραγματικά μια συνειδητοποίηση του ρόλου αυτού, να καταστούν πραγματικοί επαγγελματίες, να γίνουν ιδιοκτήτριες, να επιλέγουν την γεωργία και όχι να τους επιβάλλεται η γεωργία. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα προωθήσουμε. Και οι τοπικές αρχές επίσης. και να περάσουμε από τα κορίτσια τα οποία απλά επειδή είναι από γεωργική οικογένεια ασχολούνται με τη γεωργία να είναι κορίτσια τα οποία θα προσφέρουν καινοτομία και ανάπτυξη γιατί το επιλέγουν να σπουδάσουν ε, σε τομείς σχετικούς με τη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν τα κίνητρα τα, που θα δοθούν να είναι σημαντικά. Το TSR ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει μπορέσει να κινητοποιήσει ακόμα τις γυναίκες. Επαγγελματικοποίηση λοιπόν των γυναικών, κατάρτιση των γυναικών, πιστοτικά μέσα υπέρ των επιχειρηματιών γυναικών. Νομίζω ότι διαπιστώνουμε ότι η Γεωργία είναι ένας από τους τομείς όπου παραμένουν τεράστιες διαφορές και λείπουν τα κατάλληλα μέτρα για να καλυφθούν οι διαφορές αυτές. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και οι προλαλήσαντες, να ευχαριστώ τη Μαρίνα Πετήρ και τη Λιλιαζέρα Ροντρίγκε. Ροντρίγκες. Έκαναν εξαιρετική δουλειά οι συνεισηγήτρες όντως παρουσιάζουν πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τα προσκόμματα για τις γυναίκες ε, στην Ήπεθρο και ε, αντιμετωπίζονται διάφορα βασικά ζητήματα όπως η έλλειψη κοινωνικών ε, κρατικών υποδομών, έλλειψη πρόσβασης στην πίστη, στην, στον τεχνικό εξοπλισμό και στην ίδια τη γη που είναι βασικό εργαλείο εργασίας. Επίσης χαιρετίζω το ότι αναφέρεται και η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα είδη των κρατικών οργανώσεων και συλλόγων και ενώσεων, κυρίως για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Βεβαίως. Θα ήθελα ε, παρόλα αυτά να τονίσω ότι υπάρχουν και άλλα τέσσερα βασικά ζητήματα. Μισθολογικό χάσμα ανάμεσα ε, στις γυναίκες και στους άντρες ε, είναι κατά 10% υψηλότερο σε σχέση με άλλες περιοχές στην Ήπεθρο Για καλό θα ήταν να εκπονηθούν και επικαιροποιημένες στατιστικές για την εργασία των γυναικών στην Ήπεθρο. Δεύτερο σημείο επίσης σε πρόσβαση ε, στα γεωτεμάχια, ε, κυρίως ε, διότι σε σχέση με την εργασία που κάνουν υποτιμάται ο ρόλος τους και είναι ότι οι γυναίκες ή οι σύντροφοι των γεωκτημόνων και άρα θα πρέπει να κατοχυρωθούν περισσότερα δικαιώματα για να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, ούτως ώστε να έχουν αυτό που ονομάζουμε κοινά ε, δικαιώματα, κοινά ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Υπάρχει σε κάτι τέτοιο στο Βέλγιο. Τρίτον, θα πρέπει να αναθεωρηθούν κάποιοι ορισμοί ε, για να υπάρχουν, υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ε, στις, ε, στα δάνεια και τέταρτον διαφοροποίηση όπως άμεσο μάρκετινγκ ή αγροτουρισμός, διακοπές στο αγρόκτημα διότι αυτό μπορεί να είναι πηγή επιπρόσθετου εισοδήματος για τις γυναίκες, όχι ότι είναι δυνατόν πάντα, αλλά εάν επιθυμούν καλό θα ήταν στα πλαίσια μιας αγροτικής εκμετάλλευσης να είναι δυνατόν και να συμφιλειωθεί και η οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή στην Ήπεθρο και κυρίως αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά δεν τα υπερεύει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, όπως και προελαλήσατε, να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες ε, και εμεί χαιρετίζουμε το σχέδιο έκθεσης. Είναι όντως ποιοτική έκθεση και θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι χρειάζονται ειδικά ιδιαίτερα εξειδικευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ε, έμφυλης βίας στην Ήπεθρο. Ε, θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες γιατί υπάρχουν ζητήματα σημαντικά για την πολιτική μας ομάδα και θα θέλαμε να το τονίσουμε όπως οι, οι επιπτώσεις της κρίσης παραδείγματος χάρη για, και, ε, διότι η κρίση μας οδήγησε σε υψηλότατη ανεργία και πλήττονται κυρίως οι γυναίκες και πάλι στη Ήπεθρο. Σε πολλές περιπτώσεις επιδεινώθηκε η κατάσταση των γυναικών σε σχέση με το ρόλο τους στις οικογενειακές επιχειρήσεις θέλουμε να κατοχυρίσουμε καλύτερη πρόσβαση στη γη, στα αγροτεμάχια και θέλουμε να μιλάμε μόνο για κοινή χρήση γης, δεν θέλουμε να είναι αυτή η μοναδική βελτίωση που επιφέρουμε. Και επίσης ε, για τις μετανάστριες ε, ε, εργαζόμενες θα θέλαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν φυσικά και οι τρέχουσες ε, διαπραγματεύσεις συμφωνιών ε, ΣΕΤΑ, ΤΙΤΙΠ, ε, Μερκοσούρ και εκεί θα πρέπει να αποτυπωθεί αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα κλείνοντα να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριες και θα συνεργαστούμε για να βελτιωθεί το κείμενο. Σας ευχαριστούμε. Muchas gracias. Primero me gustaría agradecer a las... Eh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες, την κυρία Πετρή και την Ιασέα, διότι συμφωνούμε με την κατεύθυνση που παίρνει η έκθεση. Υπάρχει διάκριση εις βάρος των γυναικών στην Ήπεθρο και συνήθως οι άντρες είναι αγρότες, οι άντρες είναι αυτοί που λαμβάνουν επιδοτήσεις και οι άντρες είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για του αγρότε. Οι γυναίκε είναι αόρατες ή τουλάχιστον πολύ λιγότερο ορατέ στην γεωργία. Και εμείς λοιπόν θα υποβάλουμε τις σχετικέ τροπολογίε και θα προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε μία επιπλέον διάσταση στο θέμα, μία διάσταση που θα αφορά το υφιστάμενο μοντέλο γεωργίας, εντατική γεωργία μεγάλης κλίμακας δηλαδή κάτι το οποίο θα ενταθεί με την ε, υπογραφή συμφωνιών όπως ε, η ΣΥΤΑ για παράδειγμα και θα συνεισφέρει στην, ε, με, στην επιδείνωση των ανισοτήτων ως βάρος των γυναικών. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παρατήρουν και διονύζουν αυτές τις ανισότητες ακριβώς λόγω της δυσκολίας στην πρόσβαση των γυναικών σε διάφορες υπηρεσίες. Και ε, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το κόστος παραγωγής είναι μικρότερο, έτσι λοιπόν χρειάζεται και λιγότερο κεφάλαιο για να ασχοληθεί κανείς ε, με αυτό. Κοστίζουν πολύ λιγότερο τα ε, μέσα καλλιέργειας τα λοιπάσματα για παράδειγμα. Επίσης με την βιολογική γεωργία δεν κινδυνεύει και η υγεία των γυναικών, ιδίω η αναπαραγωγική υγεία. Αυτό το γνωρίζουμε από διάφορε μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε γυναίκες αγρότες που ασχολούνται με τι βιολογικές καλλιέργειες. Χρειάζεται λοιπόν πέραν αυτών που συζητάμε να προχωρήσουμε προς μια βιώσιμη γεωργία η οποία θα ε, συνοδεύεται και από ισότητα. Αυτό λοιπόν πιστεύουμε πως αν προωθηθεί θα επιφέρει περισσότερη ισότητα και αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε μέσω της χρηματοδότησης διαφορών έργων που θα ασχολούνται με την βιολογική γεωργία. Επίσης ε, θα επιθυμούσαμε τα λοιπάσματα και τα διάφορα ζενεκτόνα και ε, χημικά φυτοφάρμακα να αντικατασταθούν από άλλα προϊόντα τα οποία θα βλάπτουν πολύ λιγότερο το περιβάλλον και την υγεία. Και θέλουμε επίσης να προωθήσουμε ένα μοντέλο ε, γεωργίας τοπικό που οι γυναίκες θα συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Πρώτο λοιπόν μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγξουμε το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών Καλό είναι που συμπεριλαμβάνεται, αλλά αναμειγνύεται εδώ με τα θέματα των μεταφορών κτλ. Ενώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ξεχωριστό τρόπο. Να υπάρχει, θα έλεγα, μια ξεχωριστή παράγραφος γι' αυτό. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να παίξουμε τον ρόλο της βελτίωσης των υπηρεσιών. Ε, τηλεπικοινωνίες, υγεία, μεταφορές, εκπαίδευση Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο το θέμα της συλλογής των δεδομένων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για τον ρόλο των γυναικών στην Ήπεθρο, να δούμε ακριβώς ποιος είναι και ο ρόλος γενικότερα της γυναίκας στην οικολογική γεωργία. Κλείνοντας την παρέμβασή μου θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη δυνατότητα βελτίωσης των δικαιωμάτων των εργασιακών των γυναικών που απασχολούνται στη γεωργία. Ε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών στη μικροπίστωση. Ε, όλα αυτά είναι σημαντικά έτσι ώστε να έρθουν άνδρες γυναίκες στο ίδιο επίπεδο στις περιοχές της υπαίθρου. Ευχαριστώ κύριε Σελίμωβιτς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω συγχαίροντας την κυρία Πετήρ και την κυρία Σένρα για την πολύ καλή δουλειά και για την στάση την οποία έχουν κρατήσει μέχρι τώρα στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία έχει αλλάξει πάρα πολύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της γεωργίας. Η συνεισφορά όμως των γυναικών στην κοινωνία υποτιμάται συστηματικά. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες που δεν θα πρέπει να δεχόμαστε πλέον στην Ευρώπη. Υπογραμμίζουμε λοιπόν εξ αρχής την πολυλειτουργικότητα του γεωργικού τομέα, κάτι το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την παραγωγή τροφίμων, αλλά και καινοτόμες λύσεις για προϊόντα και υπηρεσίες. Όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσει η έξοδος του πληθυσμού. Λόγω ακριβώς αυτής της πολυλειτουργικότητας θα πρέπει οι γυναίκες να πάρουν ένα ρόλο πιο σημαντικό στον τομέα των του καθορισμού των πολιτικών και των στρατηγικών έτσι ώστε οι διαδικασίες λήψης απόφασης να λαμβάνονται και από την γυναικεία και από την ανδρική προοπτική. Είναι ιδιαίτερα ανδρική η εικόνα της γεωργίας σήμερα. Θα πρέπει να προωθηθεί επίσης η καινοτομία στην γεωργία και η αηφορία στη γεωργία, έτσι ώστε να είναι ελκυστικός τόπος κατοικίας των γυναικών να υπάρξει σωστή δυνατότητα εκπαίδευσης, πρόσβασης σε ε, υπηρεσίες υγείας πρώτης ποιότητας έτσι ώστε να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε όλα τα μέσα τα οποία μπορεί να θέσουμε στην διάθεση ε, των γυναικών. Να, επίσης να υπογραμμίσουμε την αποκοινού ιδιοκτησία των επιχειρήσεων των γεωργικών, την αποκοινού διαχείριση, όπως προτείνεται και στην παράγραφο 4. Θα πρέπει να τονίσουμε την προώθηση της του ε, οικολογικού σχεδιασμού και οι γυναίκε στα αγροτικέ περιοχές πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να ενισχυθεί το ρόλο του ω επιχειρηματίες και να ε, δρομολογηθεί η μετάβαση σε ε, πιο βιώσιμε και παραδοσιακέ μεθόδους ε, το οποίο θα επιφέρει προστιθέμενη αξία. Και κλείνοντα θα ήθελα να συγχαρώ τις συνεισηγήτριε για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν και να επιβεβαιώσω ότι εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες θα ε, αφούν τα σχόλια που μόλι σα έκανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Σινάντσκα έχει το λόγο στο τελευταία σκιώδη συζητήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. ακριβώ γιατί έχει ήδη γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα περιοριστώ στο περιεχόμενο της έκθεσης και θα ήθελα εδώ να συγχαρώ τις συνεισηγήτριες για κάτι που νομίζω είναι μια εξαιρετική βάση για περαιτέρω δουλειά. Οι γυναίκες της αγροτικής περιοχής δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα και η συνεισφορά τους στην κοινωνία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ε, σχετικές τροπολογίες διότι το κείμενο αφορά κυρίως την γεωργία. Ωστόσο θεωρώ πως ε, και άλλοι τομείς αξίζουν την προσοχή μας εδώ, όπως η επιχειρηματικότητα και ο τουρισμός. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι πολλές γυναίκες ε, ταξιδεύουν στις πόλεις για να εργαστούν εκεί και ε, είναι, έχουν ενεργό δράση ως ακτιβίστρες, ως πολιτικής της αγροτικές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα ήθελα να υποβάλω σχετικές τροπολογίες, καθώς και ορισμένες τροπολογίες που αφορούν τις γυναίκες με αναπηρία ή τις γυναίκες που έχουν μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία. Πιστεύω λοιπόν πως η έκθεση δεν πρέπει να παραβλέπει και αυτές τις ε, κοινωνικές ομάδες ακριβώς γιατί ε, αυτές ακριβώς οι περιοχές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Στη Σλοβακία για παράδειγμα την πατρίδα μου ε, πάσχει ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στις γυναίκες Ρωμά διότι στη Σλοβακία πολλές γυναίκες Ρωμά ζουν σε αγροτικές περιοχές και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Σε γενικές γραμμές η έκθεση είναι εξαιρετική και με χαρά αναμένω την ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Κόστιγκερ έχει το λόγο. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, συνεισηγήτριες όπως και οι προλαλήσαντες. Θεωρώ πως ε, πολλές από αυτές τις προτάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ήδη έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή Γυναικών το θέμα αυτό λίγες φορές και πιστεύω πως εδώ πρέπει να συγχαρώ την ε, δουλειά της ε, μη συνησυχήτριας. Έχει αναφερθεί σε πολλά θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την στήριξή μου σε αυτή. Είμαστε υπέρ των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές. Οι γυναίκες ε, χρειάζονται αυτή τη βελτίωση των συνθηκών και αυτό πρέπει να γίνει με ε, αύξηση των ε, μέτρων και των δράσεων που θα λαμβάνονται. Οι πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητε σε αυτά τα θέματα. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι αυτή η πολιτική, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δρέπει κουρικά σε αυτήν την πολιτική, μπορεί να κάνει συστάσεις στα κρατημέλη, να έχει συμβουλευτικό ρόλο, αλλά τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε την προσέγγισή μας, έτσι ώστε οι γυναίκες στην ε, ύπεθρο στι αγροτικές περιοχές να βοηθηθούν. Πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί οι γυναίκες στη, που ζουν στις αγροτικές περιοχές ζουν σε αυτές τις περιοχές γιατί επιλέγουν αυτή τη ζωή και να ε, βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης εκεί. Η ψηφιοποίηση για παράδειγμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα βοηθήσει τις γυναίκες εκεί να γίνουν πιο ανεξάρτητες από τις κρατικές δομές. Γι' αυτό ε, αυτή πιστεύω ψηφιοποίηση θα τους δώσει περισσότερες προοπτικές. Επίσης μπορούμε να αντλήσουμε κονδύλια από διάφορα ταμεία, ταμεία πούμε, για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου και να στοχεύσουμε σε αυτές τις ομάδες γυναικών, να ε, στοχεύσουμε έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, να βελτιωθούν και να αυξηθούν οι επενδύσεις και πολλά άλλα ακόμα που θα βοηθήσουν τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές. Θεωρώ πως ε, η έκθεση αυτή δεν ε, αφορά μόνο ε, αυτόν τον στενό ρόλο των γυναικών, αφορά πολλά περισσότερα και τα οποία πρέπει να αναφερθούν. Και επίσης να πω πως δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο στα αρνητικά στοιχεία, διότι έτσι δεν προχωράμε παραπέρα. Πρέπει να αναφερθούμε στις δυνατότητε που έχουμε, στις ευκαιρίε που έχουν οι γυναίκες για να βελτιώσουν την ε, ζωή τους και τη θέση τους εκεί. Πρέπει επίσης να ε, συνυπολογίσουμε την καινοτομία στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις ε, που ασχολούνται με τη γεωργία. Ε, εδώ βέβαια η εθνική νομοθεσία είναι ε, περισσότερο αρμόδια από εμά. Υπάρχει το, ε, το σχετικό δίκαιο, γι' αυτό πρέπει να δούμε και αυτήν την άποψη. Να πω κλείνοντας πως υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγνιου έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Κώστινγκερ είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών πολλά από αυτά με τα οποία ασχολούμαστε. Η κατοχή γης, για παράδειγμα. Και εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα στα κρατη Και είναι προφανές ότι τα κράτη-μέλη επενδύουν πολύ στην ε, Γεωργία και σίγουρα πολλές γυναίκες δραστηριοποιούνται εκεί. Ο κύριος Ταραμπέλα νομίζω αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα στη Γεωργία ανάμεσα σε άντρε και γυναίκε. Εγώ να πω ότι στη δική μου χώρα ε, έχουν γίνει τόσα πολλά που δεν αναγνωρίζω ε, την πατρίδα μου. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμω πιστεύω πως αυτό δεν έγινε χωρίς λόγο. Άλλαξε για παράδειγμα το βάρος των σάκων με τα ε, τρόφιμα. Κάποτε τα τρόφιμα τα μετέφεραν σε σακιά που ζύγιζαν 100 κιλά το καθένα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν μια γυναίκα να μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Άλλαξαν λοιπόν τα πράγματα και γι' αυτό οι άντρε που μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το βάρος δούλευαν σε αυτό αυτές ε, τις ε, δουλειές, πληρώνονταν περισσότερο. Αυτό δεν έχει να κάνει με ε, ισότητα, αυτό έχει να κάνει με απλά μαθηματικά. Τώρα, αναφέρθηκε το ότι πρέπει να δοθούν χρήματα αποκλειστικά σε γυναίκες από κοινοτικά ταμεία. Αυτό λοιπόν θεωρώ πως αποτελεί παράδειγμα διακρίσεων εις βάρος αντίθετα των ανδρών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε όταν πάμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να μην γίνεται διάκριση βάρος των ανδρών. Ας ε, δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα, ίσως λίγο τραβηγμένο. Μία γυναίκα για παράδειγμα κληρονομεί μία μεγάλη έκταση ε, γης κάνει αίτηση για επιχορήγηση και την παίρνει. Και μια γυναίκα λοιπόν που έχει 5.000 εκτάρια γη στην κατοχή της και ένας άνδρας που νοικιάζει, ε, 50 εκτάρια ε, γης κάνει την ίδια αίτηση και απορρίπτεται αυτή. Αυτό λοιπόν είναι ε, διάκριση. Επίσης να πούμε πως ε, η γεωργία δεν είναι επάγγελμα. Η γεωργία αφορά και το εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν Πιστεύω πως ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην παραπλανούμε στους ορισμούς. Υπάρχουν διάφορα επαγγέλματα, συμβουλευτικές δραστηριότητες για παράδειγμα, χρηματοοικονομικά, αυτά είναι επαγγέλματα. Η ε, γεωργία όμως είναι τέχνη, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι δουλειά. Thank you very uh, uh, Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Το θέμα είναι να μην μείνουμε στα λόγια. Υπάρχουν πολλά θέματα. Δυστυχώς, όπως είπαν και διάφοροι ομιλητές, πολλά από αυτά τα θέματα είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο όμως είναι εντός είναι η λιτότητα η φιλική στάση απέναντι στα πιστοτικά ιδρύματα και η αντίληψη η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε με ευτήρια στις γεωργικές περιοχές. Το δικό μου county δεν έχει πλέον με ευτήριο, το ίδιο ισχύει και για το γειτονικό. Όταν είσαι γυναίκα λοιπόν καλό είναι αν θες να γεννήσεις να είσαι κοντά σε τέτοιου είδους νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει δυόμιση ώρες αυτοκίνητο για μένα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί υπέρ των γυναικών. Τελικά οι άνθρωποι θέλουν, λέγεται, να φεύγουν από τις γεωργικές περιοχές. Όχι, δεν ήθελαν να φεύγουν. Ε, αναγκάστηκαν να φύγουν. Και πώς μπορεί να περιμένει κανείς από ανθρώπους χωρίς τις βασικές υπηρεσίες ε, να μένουν στις περιοχές αυτές. Βέβαια, αν όλα τα χρήματά αυτά δίνει στις τράπεζες, ε, τότε τα νοσοκομεία τι να μείνει γι' αυτό. Ο κύριος Ντές, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω τις συνεισηγήτριες εκ μέρους της δικής μου πολιτικής ομάδας και να αναφερθώ σε κάτι που είπε και η κυρία Κιώστινγκερ παρατηρούμε πολύ διαφορετικές ε, καταστάσεις ανάλογα με την περιοχή. Βλέπουμε πολλά διαφορετικά μοντέλα στην Ευρώπη ε, που ε, έχουν άμεσα να κάνουν με τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Στη δεκαετία του 80 ήμουν στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και ήμουν ανάμεσα στους βουλευτές που δούλεψαν ε, γεωργική νομοθεσία. Είδαμε λοιπόν ε, πως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα μιας υποχρεωτικής ε, ασφάλισης για τους αγρότες, άντρες και γυναίκες. Αυτό βέβαια συνεπα... συνεπαγόταν ότι έπρεπε να πληρώσουν και υποχρεωτικές εισφορές ε, τώρα, έχει τύχει να μιλήσω με γυναίκες οι οποίες τότε στη δεκαετία του 80 είχαν εκφράσει παράπονα για το ότι έπρεπε υποχρεωτικά να πληρώνουν εισφορές ε, και ξέρετε τι μου είπαν, με ευχαρίστησαν γιατί τώρα έχουν σύνταξη και μπορούν να ζήσουν από αυτή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές να ε, στηρίζονται. Τώρα, κάτι άλλο ε, που αφορά την, ε, τις αγροτικές περιοχές στην Ήπεθρο είναι και οι διαφορές που αναφέρα πιο πριν. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ε, ας δείτε τη Βαβαρία, για παράδειγμα. στη Βαβαρία, που είναι μια κυρίως αγροτική περιοχή, έχουμε 1,7% ανεργία. Πολύ χαμηλή. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να δούμε τις διαφορές όχι μόνο ανά κράτος αλλά και ανά περιοχή και ε, δεν πρέπει να κατηγορούμε συνέχεια τις Βρυξέλλες στην Ευρώπη αλλά να βλέπουμε και τι καλό έχει κάνει που στην προκειμένη περίπτωση έχει στηρίξει πάρα πολύ τις αγροτικές ε, περιοχές ιδιαίτερα ε, μάλιστα βοηθώντας τις γυναίκες να δραστηριοποιούνται και να διαβιώνουν αξιοπρεπώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. <clears throat> Νομίζω ότι έχουν ήδη τεθεί τα περισσότερα από τα θέματα από τις προηγούμενες ομιλίες. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε τη σωστή διάγνωση για τη θέση των γυναικών στην γεωργία. Προφανώς και μπορεί να υπάρξουν προφανείς αλλαγές και προφανώς υπάρχουν και σημαντικές διαφορές από τη μία περιοχή στην άλλη. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά όπως ο συνδυασμός της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, το pay gap, η διαφορά στις αμοιβέ, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υπέρ του πληθυσμού και θα πρέπει λοιπόν μέσω της σωστής διάγνωσης να κατανοήσουμε ποια είναι η κατάσταση των γυναικών στην Ήπεθρο σήμερα sobre la cuestión competencial y creo Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο ε, αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών οργάνων. Υπάρχει ένα θέμα εδώ αρμοδιοτήτων και να πούμε όμως ότι η ισότητα ανδρών γυναικών είναι μια βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιείται η πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και με μια έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορέσουμε να κάνουμε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες να προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το νομοθετικό κομμάτι το οποίο μας ανήκει έτσι ώστε να κάνουμε τις απαιτούμενες συστάσεις στα κράτη-μέλη για τις πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν την ζωή των γυναικών στην Ήπεθρο. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς την σωστή κατεύθυνση και μέσω των τροπολογιών μας. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Συνεπώς θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ε, εφόσον το επιθυμεί βέβαια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά τα οποία μέχρι τώρα υπόθηκαν. Οι δύο εκθέσεις ήταν εξαιρετικές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις θέσεις της σε πολλά από τα θέματα τα οποία έχουν ήδη υπογραμμιστεί. Νομίζω ότι έχουμε κάποια μέσα τα οποία μπορεί να είναι αποτελεσματικά εφόσον τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες το επιθυμούν. Είναι λοιπόν πολύ σωστό που επισύρεται την προσοχή των περιφερειών στα θέματα της ανάπτυξης της υπαίθρου και στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις γεωργικές περιοχές, έτσι ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές οι επενδύσεις σαν παράδειγμα στις βασικές υπηρεσίες, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη για την ανάπτυξη των γεωργικών επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, στις οποίες είναι σημαντική η παρουσία των γυναικών. Είναι στόχοι που μπορούν να επιδιωχθούν με αρκετή ευκολία στα πλαίσια της πολιτικής για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι έχω ένα όνειρο εδώ, να βελτιωθούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων στην Γεωργία και στην Ήπεθρο. Η ψηφιοποίηση μπορεί να αλλάξει και να αυξήσει τις δυνατότητες που παρέχονται στις γυναίκες στις γεωργικές περιοχές. Και εδώ θα πρέπει να σπρώξουμε. Να πω επίσης ότι τα οικονομικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων ε, των, ε, του, σαν παράδειγμα της έλλειψης πιστώσεων ε, μπορούμε να παίξουμε και εκεί έναν κάποιο σημαντικό θα έλεγα ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω τώρα από την κυρία Σέντρα να πάρει το λόγο. Bueno, pues creo que Δεν έχω πάρα πολλά να πω πια εδώ. Να πω ότι ήταν ικανοποιητική η συζήτηση, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη μεγάλη συμμετοχή να πω ότι υπήρχαν ορισμένες πλευρές της έκθεσης τις οποίες ε, συμμερίζομαι, κάποιες άλλες που μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο. Να ελπίσω ότι θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες και πολλές ε, συνεισφορές έτσι ώστε το έγγραφο αυτό να βελτιωθεί επιπλέον. Πετήρα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και εκ των προτέρων αυτούς που θα καταθέσουν τροπολογίες. Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη Υπέθρου υπάρχει ένα υποπρόγραμμα για τις γυναίκες στην Ήπεθρο, το οποίο όμως δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα από τα κράτη-μέλη. Επειδή κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στη χρήση του προγράμματο, θέλω να σχολιάσω το ότι η μη διακριτική μεταχείριση και η ισότητα είναι οι δύο προϋποθέσεις για το πρόγραμμα αυτό. Και επειδή ακριβώς συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, δεν θα πλήξει αυτό του άντρε στην Ήπεθρο αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Ακούσαμε επίσης κάποιες ε, παρατηρήσεις για το θέμα της αρμοδιότητας. Για το θε... Ως προς το ζήτημα της επικουρικότητας, εντοπίσαμε κάποιες δυσκολίες και είναι σαφές ότι όταν αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους δυσκολίες είναι χρήσιμο να τις φέρνουμε στην επιφάνεια. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουν υπάρξει επίσης και ορισμένες ε, τροπολογίες οι οποίες ε, θα έλεγα υπερβαίνουν το πλαίσιο της ε, συγκεκριμένης πρότασης. Αν αρχίσουμε να πλαταίνουμε ιδιαίτερα και ασχολούμεθα με θέματα εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα στις διάφορες χώρες και με άλλα θέματα όπως η οικολογία, η βιολογική, η οργανική γεωργία κτλ. Τότε σε αυτή την περίπτωση έχω την εντύπωση ότι διακινδυνεύουμε την φύση της συγκεκριμένης έκθεσης και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μείνουμε στις βασικές αρμοδιότητες των δύο επιτροπών. Σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις ε, συνεισηγήτριες. Σας ευχαριστώ για τις ε, συζητήσεις μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο παρελθόν. Έχουμε καταπολεμήσει τη διακριτική μεταχείριση. Έχουμε πετύχει πράγματα στον τομέα της ισότητας. Κινητοποιούμαστε για τα εκκρεμή προβλήματα. Ε, είναι προεξάρουσα η θέση των αντρών. Ε, ξέρετε, αυτό συνδέεται και με την ίδια τη φύση του επαγγέλματος οι γυναίκες. συχνά δεν ασχολούνται με τις αμυγός ε, γεωργικές υπηρεσίες. Εξασφαλίζουν κάποιες υπηρεσίες ένα επιπρόσθετο εισόδημα. Νομίζω ότι είναι αλληλοσυμπληρούμενες αυτές οι δραστηριότητες. Επίσης η ψηφιοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει αλλάξει πολύ κατάσταση. Εγώ θυμάμαι πριν από 40-50 χρόνια πώς ήταν αναγκασμένη να δουλεύει η γυναίκα, η, συγγνώμη, η μητέρα μου. Φυσικά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Όντως θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω προέδοδος, όντως θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στην παιδεία, στην κατάρτιση, στη δανειοδότηση. Κλείνοντας, θέλω να σα πω ότι η 14η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τι τροπολογίε. Το Φεβρουάριο πάνω κάτω νομίζω μπορούμε να προβλέψουμε την έγκριση αυτή τη νομοδότησης. Σα ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε για την ε, μεικτή συνεδρίαση. Νομίζω ότι από κοινού μπορούμε πολλά να καταφέρουμε.